Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, κυρίες και κύριοι. Ενώπιόν μας έχουμε πέντε πολύ απαιτητικά χρόνια για τα οποία είμαι πεπισμένη ότι θα είναι κρίσιμη σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κρίση είχε καταστροφικές συνέπειες σε πολλές χώρες. Η ανεργία των νέων έχει φτάσει σε απαράδεκτα επίπεδα σε πολλές περιοχές της Ευρώπης η πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι η εξή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αντιμετωπίσει τις ανάγκες των λαών τα επόμενα πέντε χρόνια θα είναι κρίσιμα στην αποκατάσταση εμπιστοσύνης απέναντι σε αυτό το θεσμικό όργανο. Γι' αυτό έχουμε ε, πρέπει να κάνουμε το θεματολόγιο για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατική αλλαγή να επιτύχει. Αυτό το θεματολόγιο θα εφαρμοστεί από μια ισχυρή ομάδα μέσω αμοιβαία συνεργασία. Σε αυτή την αμοιβαία συνεργασία βλέπω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως έναν από τους εταίρους κλειδί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέλω να δεσμευτώ ότι θα καταβάλω κάθε προσπάθεια να ενισχύσω τη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Επιτροπής. Ως πρώην Πρωθυπουργό και μέλος του Κοινοβουλίου βεβαίως εκτιμώ τη σημασία του συνεισφοράς του Κοινοβουλίου στην εξέβρεση λύσεων και βεβαίως την υλοποίηση της κοινή ατζέντα για προς των Ευρωπαίων πολιτών. Λοιπόν, αγαπητά μέλη, είναι τιμή για μένα και έρχομαι με μεγάλη ταπεινοφροσύνη για να καθίσω ενώπιόν σας ε, ω υποψήφια για τη θέση της Αντιπροέδρου για την Ενεργειακή Ένωση. Η πατρίδα μου η Σλοβενία εντάχθηκε στην ευρωπαϊκή οικογένεια πριν από 10 χρόνια. Για μένα αυτό ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Εγώ και η γενιά μου γνωρίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο χώρος στον οποίο ανήκουμε. Αποτελεί λύση, δεν είναι πρόβλημα. Και η δημιουργία μιας ενεργειακής ένωσης με την σύγκληση των κρατών μελών στον τομέα της ενέργειας και των πολιτικών για το κλίμα έχει κάθε δυνατότητα να αποτελέσει ε, έναν ένα βήμα προς την στρατηγική της Ευρώπης για να ξεπεραστεί η κρίση. Αυτό ακριβώς είπε ο πρόεδρος Γιούνκερ όταν απευθύνθηκε στο Κοινοβούλιο και αυτό είναι και το όραμά μου. Η εξασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας, της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στην παγκόσμια αγορά και η ενίσχυση μιας βιώσιμης πράσινης ανάπτυξης με βάση ξεκάθαρους στόχους για το κλίμα, όπως επίσης ε, ε, και άλλοι, άλλοι στόχοι που αποτελούν τις βασικές προκλήσεις της εποχής μας. Ως μέλος ε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που μέχρι πρόσφατα, έχω πλήρη συνέστηση το πόσο σύνθετα είναι τα θέματα της ενέργειας. Όχι μόνο έπαιξα ενεργό ρόλο ε, στη στρατηγική των συζητήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά ήμουν απολύτως προσιλωμένη στην υλοποίηση των απαραίτητων μέτρων σε εθνικό επίπεδο. Μεταξύ άλλων είμαι περήφανη να πω ότι κατά τη διάρκεια της Πρωθυπουργία μου στη Σλοβενία μπορέσαμε να υλοποιήσουμε το τρίτο ενεργειακό πακέτο. Κυρίες και κύριοι, ε, ανέλαβα Πρωθυπουργό σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους στην ιστορία του νεαρού μας κράτου και ε, πραγματικά μέσω μιας σωστά μετρημένης και συνεπούς πολιτικής με βάση τις ευρωπαϊκές αρχές και τις δεσμεύσεις μας καταφέραμε να βγάλουμε τη Σλοβενία από την χειρότερη οικονομική κρίση. Πιστέψτε με, είμαι συνηθισμένη να δουλεύω σε συνθήκες υψηλού στρες, επίσης όμως γνωρίζω ότι το άγγιγμα της γυναίκας καμιά φορά μπορεί να ηρεμεί τα πράγματα. Θα ήθελα τώρα να πω δύο λόγια για τον ορισμό μου ως επιτρόπο. Όπως θα γνωρίζετε ε, υπήρχε μια προθεσμία υποβολή των ονομάτων των υποψηφίων και αυτή ήταν το τέλο Ιουλίου. Δεδομένου ότι δεν μπορούσε να επιτεθεί συμφωνία ανάμεσα στου εταίρου του συνασπισμού, ε, και δεν υπήρχε ένας ε, υποψήφιος, είχαμε δύο δυνατότητες. Είτε να μην στείλουμε κανένα όνομα στις Βρυξέλλες και να περιμένουμε τη νέα κυβέρνηση να το κάνει στο τέλος Σεπτεμβρίου και όλοι φαντάζεστε τι επιπτώσεις θα είχε αυτό στην Επιτροπή ή να στείλουμε έναν κατάλογο ονομάτων. Αυτός ο κατάλογος αποτελείται από τρία ονόματα, συμπεριλαμβανομένοι και του δικού μου και την τελική απόφαση την έλαβε ο πρόεδρος Γιούγκερ. Αυτά συνέβησαν και τίποτε άλλο. Θα ήθελα τώρα να στραφώ στην κοινή μας πρόκληση, τη δημιουργία της Ενεργειακής Ένωσης. Η πατρίδα μου δεν είναι η μόνη χώρα μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία λόγω της γεωγραφικής της θέσης ε, αντιμετωπίζει κινδύνους στην ενεργειακή ασφάλεια όπως μια, την υπερβολική εξάρτηση από έναν μη Ευρω... κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης προμηθευτή. Έτσι λοιπόν δεν χρειάζεται να, με... πιστώ ότι κανένα κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις ενεργειακές δυσκολίες από μόνος του. Οι ενεργειακές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν απαιτούν τώρα περισσότερο από ποτέ μια ισχυρή ενωμένη Ευρώπη που θα μιλά με μια φωνή διεθνώς και, και μια καλά λειτουργούσα εσωτερική αγορά ενέργειας. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει 53% της ενέργειάς της. αυτά τα νούμερα είναι πάρα πολύ σημαντικά για να καταλάβουμε τη σημασία του έργου της, Ευρωπα... της ε, ε, Ενεργειακής Ένωσης. Καθημερινά εισάγουμε ενέργεια αξίας 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Το 2013 το κόστος της ενέργειας έφτασε 400 δισεκατομμύρια ευρώ και ήταν το 1 πέμπτο του συνόλου των εισαγωγών μας. Η εξάρτηση από τις εισαγωγές από μόνη αποτελεί κίνδυνο, αλλά όταν αυτό συνδυάζεται με εξάρτηση από έναν μοναδικό εταίρο, τα πράγματα μπορεί να ξεφύγουν. Το γεγονός ότι έξι κράτη-μέλη ε, στηρίζονται αποκλειστικά σε, σε μια ξένη πηγή για την προμήθεια αερίου, ενώ πολλά άλλα έχουν έκθεση που ξεπερνά το 60% είναι γεγονός. Τα νούμερα αυτά μας δείχνουν πόσο σημαντικό είναι το όραμά μας. Το όραμα μιας ε, των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία θα συμπτύξουν μια ανθεκτική ε, ενεργειακή ένωση το όραμά μου είναι μια ανθεκτική ενεργειακή ένωση η οποία θα, έχει, θα βλέπει στο μέλλον σε, σχέση με την κλιματική αλλαγή η οποία θα στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες. Πρώτον, η ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς και αύξηση της ασφάλειας ε, της, ενέργεια, της προμήθειας ενέργειας μέσω της διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας και με την ε, διασύνδεση της ε, υποδομής με τους συνδετήριους αγωγούς, όπως επίσης και μια ενωμένη παρουσία στις διεθνείς ενεργειακές αγορές. Δεύτερον, να συνεχίσουμε να προωθούμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διευρύνοντας την, ε, και ενισχύοντας την ευρωπαϊκή κυριαρχία στην τεχνολογία, έρευνα και ανάπτυξη μέσω πρωτοβουλειών ε, για τις επενδύσεις, την προώθηση της ε, ευαισθητοποίησης. Τρίτον, η ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της πράσινης ανάπτυξης με τη διατήρηση της κυρίαρχης θέσης στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την επίτευξη των στόχων του 2020 και, την, και τους φιλόδοξους στόχους για το 2030 ε, σε σχέση με τα κίνητρα που θα μειώσουν την ενεργειακή κατανάλωση και θα αυξήσουν την αποδοτικότητα της ενέργειας. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι από όπως βλέπουμε τα πράγματα σήμερα μπορεί να μοιάζει ότι η σχέση μας με τη Ρωσία είναι το κρίσιμο ζήτημα για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, βραχυπρόθεσμα, η ασφάλεια της προμήθειας αερίου οπωσδήποτε είναι ένα θέμα που πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα. Αλλά δεν θα πρέπει να σταματήσουμε εδώ, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν και άλλοι μακροπρόθεσμοι κίνδυνοι που πρέπει να αντιμετωπιστούν για την Ευρώπη και τους πολίτες στον τομέα της ενέργειας. Η επίτευξη των κλιματικών στόχων μας, ενώ ταυτόχρονα η ενίσχυση τη ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας πρέπει να παραμείνει πρώτη προτεραιότητα της ατζέντα μας. Είμαι πεπισμένη ότι ε, τον, αν κάνουμε την, εσωτερική ενεργειακή αγορά μία πραγματικότητα χωρίς επιστροφή και αν ε, εφαρμόσουμε τις, ε, τους κλιματικούς στόχους που έχουν συμφωνηθεί ξεκινώντας από το πακέτο 2020 σε συνδυασμό με ένα μεγάλο πακέτο επενδύσεων, εκτεταμένων επενδύσεων όπως ανακοίνωσε ο κύριος Γιούνκερ θα έχουμε το κλειδί για να αντιμετωπίσουμε σωστά και την οικονομική και την κλιματική αλλαγή και τις δυσκολίες της εποχής μας. Μόνο επίσπευση των επενδύσεων στην ενεργειακή υποδομή, καθαρές ε, τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον και κυρίως από δοτική χρήση της ενέργειας μπορούν να μας βοηθήσουν να ξεπεράσουμε το πρόβλημα. Ε, το ενεργειακό πλαίσιο του 2030 πρέπει να μας καθοδηγεί. Κυρίες και κύριοι, αυτό φυσικά θα απαιτήσει και χρόνο και σκληρή δουλειά και απαιτείται συνεργασία ανάμεσα στα θεσμικά όργανα. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι είμαι απολύτως προσιλωμένη στη συνεργασία με το Κοινοβούλιο και τις Επιτροπές Ήτρε και Ένβη. Θα ήθελα να αναλύσουμε τις αλλαγές, τις δυσκολίες από κοινού, να αποφασίσουμε για συγκεκριμένες δράσεις και τις φιλοδοξίες για την εφαρμογή της Ενεργειακής Ένωσης και τους στόχους της κλιματικής αλλαγής. Αυτό θα μας ε, θα φέρει την αλλαγή. Η αλλαγή που χρειαζόμαστε για να ενισχύσουμε την οικονομική ανάπτυξη, νέε θέσει εργασία, ενώ θα μειωθεί η κατανάλωση ενέργεια και θα ενισχυθεί η ενεργειακή ασφάλεια. Στο παρελθόν η Ευρώπη έχει δείξει ότι είναι δυνατόν να επιτευχθεί οικονομική ανάπτυξη και μείωση τη κατανάλωση ενέργεια ταυτόχρονα. Αλλά πρέπει να προχωρήσουμε περισσότερα και να το γνωρίζουν αυτό και οι πολίτε μα. Εάν θεωρήσουμε ότι το 50% τη ενέργεια ενέργειας χρησιμοποιείται για θέρμανση ψήξη, είναι προφανές ότι η δυνατότητα για εξοικονόμηση δεν έχει εξαντληθεί. Εδώ μπορούμε να πετύχουμε ταυτόχρονα δύο πράγματα. Η, ανανέωση, ενεργειακή ανανέωση των κτηρίων με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ενώ ταυτόχρονα θα, μειώνεται η θα μειώνονται οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και η εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις εισαγωγές. Αυτό είναι ένα είδος βιώσιμης ανάπτυξης που χρειάζεται η Ευρώπη. Θα καταβάλω κάθε προσπάθεια έτσι ώστε ένα σημαντικό κομμάτι των 300 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα επενδυθούν και τα οποία ανακοίνωσε ο πρόεδρος Γιούνκερ στην εναρκτήρια ομιλία του να δοθεί προς έργα ενεργειακής απόδοσης που θα ενισχύσουν την πράσινη ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ευρώπη. Αυτό είναι ο σωστός δρόμος για την Ευρώπη. Η επίτευξη αυτών των στόχων θα απαιτήσει πραγματικά ομαδική δουλειά και συγκέντρωση ε, σε συγκεκριμένα έργα μεγάλης σημασίας. Επίσης από την πλευρά της Επιτροπής ε, στο πλαίσιο της, του θεματολογίου για τις θέσεις εργασίας, την ανάπτυξη, τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατική αλλαγή θα αναλάβω ενεργό ρόλο για τις δύο ε, βασικές προτεραιότητες. Θα συντονίσω και θα καθοδηγήσω τη δουλειά με τους ε, συναδέλφους επιτρόπους που, ε, αφορούν και που έχουν σχέση με την Ενεργειακή Ένωση. Θα είναι ε, καθήκον μου να εξασφαλίσω ότι οι ιδέες και λύσεις από, τη, από τους συγκεκριμένους τομείς να ενσωματωθούν στρατηγικά σε μια πραγματικά καλά συντονισμένη δράση. Μία ακόμα πρόταση, αν αγαπητά μέλη των Επιτροπών, σας ευχαριστώ για την